Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz. Bitte schnell, συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Ισχέ η πολιτική της Ρωσίας στον τομέα της ε, ενέργειας και του εμπορίου ως πολιτικό όπλο κατά των ε, γειτόνων της, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά της Ουκρανίας, αλλά όχι μόνο κατά της ε, Ουκρανίας. Οι δηλώσεις που γίνονται στη Μόσχα και τα μέτρα που λαμβάνονται Νομίζω το είπα και σε μια δήλωση τύπου μαζί με τον συνάδελφο Σάρος Βόλσκι. Αυτά λοιπόν όλα καταδεικνύουν μια κατάσταση που είναι απαράδεκτη για μια ελεύθερη Ευρώπη. Η συμφωνία του Ελσίνκη της δεκαετίας ε, του 70 ε, έχει υπογραφεί και δεσμεύει και τη Ρωσία και ισχύει ακόμη. Και εκεί λέγεται ότι κάθε κράτος στην Ευρώπη πρέπει να λαμβάνει ελεύθερα την απόφαση για την κατεύθυνσή του, για τις σχέσεις με τις άλλες χώρες, για συμμαχίες, συμφωνίες, εταιρικέ σχέσεις. Ο καθένας μπορεί να λάβει οποιασδήποτε αποφάσεις επιθυμεί. Αυτή είναι ε, υποχρέωση δημοσίου δικαίου, συμβατική όλων των χωρών της Ευρώπης και τα μέτρα που έλαβε η Ρωσία θεωρώ ότι είναι παραβίαση της συμφωνίας του Ελσίνκη και υπενθυμίζω ότι παραβιάζονται και κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου από τη Ρωσία. Είναι απαράδεκτο. Όταν μια χώρα θέλει να συνάψει ε, στενότερη σχέση με κάποια άλλη, να έχει προβλήματα με τη Ρωσία. Δεν είναι ε, ε επίσης προς το συμφέρον μας να είναι κακές οι σχέσεις μεταξύ της ε, Ουκρανίας και της Ρωσίας. Είναι καλό να μην υπάρχουν εντάσεις στην Ευρώπη, να μην υπάρχουν παγωμένες σειράξει σε διάφορα τμήματα της Ευρώπης. Όλα αυτά δεν βοηθούν την Ευρώπη που θέλουμε. Πώς θα διαμορφώσει τις ε, σχέσεις της ε, μία χώρα, όπως η Ουκρανία, είναι ε, δικαίωμα κάθε χώρας. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει τη θέλησή του ούτε από τις Βρυξέλλες ούτε από τη Μόσχα. Πρέπει να αποφασίζεται για την Ουκρανία στο Κίεβο. Ούτε στη Ρωσία ούτε στη Μόσχα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι σωστές ε, προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτό και η απόφαση των Υπουργών το 12, το Δεκέμβριο του 12, ε, ε, ε, κατά την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής του Βίλνιους πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν και οι αποφάσεις, η απόφαση για το ποιος θα, για το αν το Κίεβο θα ε, ε, ε, συμμετάσχει σε αυτές τις αποφάσεις είναι θέμα Κιέβου. Μην ξεκινήσουμε όμως συζήτηση για, για όλο το θέμα της συνοδοκορφής στη Βίλνα και την Συμφωνία Σύμβασης. Θα συζητήσουμε την έκθεση Βόλσκι ε, το προτιμάζουν οι συνάδελφοι και θα το έχουμε άλλες περιστάσεις στη διάθεσή μας ε, για να συζητήσουμε σχετικά με την σύνοδο στη Βίλνα. Και τι πρόοδοι έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Σήμερα θα πρέπει να περάσουμε ένα καθαρό μήνυμα που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Και χαίρομαι που έχουμε εδώ ανάμεσά μας τον Ουκρανό πρέσβη και ο Τσέναφος Βίγκας από τη δική μας πλευρά είναι αυτά τα θέματα. Ας έχουμε τοποθετήσει μια σύντομη μετά συζήτηση και κατά τις 12 θα τελειώσω αυτό το σημείο και θα σας ζητήσω να κάνουμε και ένα άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης η Κλίσκο και η από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης θα μας παρουσιάσουν ε, την ε, θέση τους. Δεν μπόρεσαν να έρθουν τον Ιούνιο διότι ε, απασχολούνταν σε μια συνεδρίαση της Ουκρανικής Βολή. Και θα τους καλωσορίσω και αυτούς. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο και παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που αμελητεί την πρώτη μέρα εργασία σα μετά τις καλοκαιρινές εκοπές κάνετε αυτή τη συζήτηση για το θέμα σας. Ήταν πολύ γεμάτο αυτό το καλοκαίρι. Προσπάθησε η Ουκρανία να κάνει όλες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την συμφωνία σύνδεση που θέλουν υπογραφεί στη Βίνα Και μια από τις κύριες εξελίξεις τις οποίες ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να κάνει με το νομοσχέδιο σχετικά με τις ε, διώξει Παρόλα τα όσα κάναμε όμως είδαμε ότι υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να επιβιδίσει η Ουκρανία και θα ήθελα εδώ να δηλώσουμε στεναρός ότι πέρα από ε, τις προσπάθειες να μας τρομάξουν θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία σύνδεσής μας τον Νοέμβριο. Η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμετάκλητη. Πριν από δύο εβδομάδες η τηλεονική αρχή της, της ε, Ρωσίας πέρασε σχεδόν όλους τους Ουκρανούς εξαγωγούς ε, στην κατηγορία κινδύνου στο σύστημά τους. Στην ουσία σημαίνει ότι μπλοκαρίστηκαν εξαγωγές μας τη Ρωσία ε, διάφορη λεπτομερή υποχρεωτική έλεγχη για όλα τα προϊόντα σχεδόν από την Ουκρανία ε, εφαρμόζονται πλέον για βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Οι επιχειρήσει μα που στοχοθετούνται από αυτέ τι δράσει προσωπεύουν τα δύο τρίτα τη οικονομία μα, Η βαριά βιομηχανία, τα, η που σημαίνουν ε, χιλιάδε θέσει εργασία. Ήταν όμω στεναρή και σοβαρή η κυβέρνησή μα, στο ότι θα πρέπει σε επαφέ με την Ρωσία ε, να έχουμε ε, μία λύση αυτών των θεμάτων. Μετά από συναντήσεις των Προέδρων μας, μια κυβερνητική ε, αντιπροσωπεία μας με επικεφαλής του Υπουργό μας πήγε στη Μόσχα την Δευτέρα και είχαν, είχε ένα πακέτο επικοδομικών προτάσεων για να υπάρξει λύση δεδομένου ότι θα γίνει υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσής μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε όλους τους παρέτητους μηχανισμούς για να βρούμε τις λύσεις. Ε, ε, ε, να βρούμε τους, τους εταίρους μας. Και άρα λοιπόν αυτό το δηλώσαμε στον κύριο Κλάσιο, τον εκπρόσωπο Πούτιν, αλλά αυτός δήλωσε ότι θα σταματήσει να είναι στρατηγικός εταίρος η Ουκρανία για μας, ούτε καν θα θεωρούμε ότι είναι μέρος του διεθνούς ε, δικαίου. Θα θεωρούμε ότι είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα είπε η Μόσχα ότι θα επαναφέρει ειδικού μηχανισμούς και λόγω να υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Παραδείγματο χάρη ενιαίε κατηγορίε για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την Ουκρανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλλον αυτό θα το αντιμετωπίσουμε μετά την επιτυχία που σίγουρα θα έχουμε στην Βίλνα και φυσικά όλες αυτές οι δράσεις της Μόσχας ε, βλάπτουν τους πάντες ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και την ίδια τη Ρωσία. Αυτή τη στρατηγική την εφαρμόζει η Ρωσία παρόλο που έχει δεσμευθεί να μην χρησιμοποιήσει οικονομική πίεση για να επιβάλλει τα δικά της συμφέροντα στην Ουκρανία και να βλάψει την εθνική μας ε, κυριαρχία. Αυτό το είχε συμφωνήσει στο μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994 τότε που είχε μπει η Ουκρανία στην θήκη μη εξάπλωση ε, των, ε, των ατομικών όπλων. Θα ήθελα να εκφράσω σε εσά την εκτίμησή μα για, τα, ε, για τις δηλώσεις που έκαναν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου από όλε τι μεγάλε πολιτικέ ομάδε που δείχνουν ότι είναι δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ ημών. Εκτιμούμε και τα σχόλια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έψεξε τη Μόσχα για αυτή τη συμπεριφορά, ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη. Σε αυτή τις συνθήκες όμως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο από δηλώσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι συνδυασμός πολιτικής και ηθικής στήριξης προς τη χώρα μου. Πρώτον, αυτές τις μέρες χρειάζεται η Ουκρανία όλες οι πολιτικές οικογένειες του Ευρωκοινοβουλίου να συνυπογράψουν ε, ε, το ότι θέλουν την συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρατία. Μετά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακοινώσει μια τελική απόφαση των κρατών μελών σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής της 21 Οκτωβρίου και όποτε να μην γίνει ε, αναβολή της συμφωνίας που μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά θα πρέπει να γίνει γρήγορη εφαρμογή της συμφωνίας μόνο εφόσον αυτό το δεχτεί το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να βασιζόμαστε στη στήριξή σας, να συμφωνήσετε επ' αυτού αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Τέταρτον, θα πρέπει να εντακοποιήσουμε τις επαφές ανάμεσα στην ηγεσία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, των κρατών μελών, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Πέμπτον, θα πρέπει επίσης να ξεκινήσουμε μία εκστρατεία πληροφόρηση σχετικά με τα προνόμια που θα φέρει αυτή η συμφωνία σύνδεσης και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Από δημοκρατική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική άποψη. Έκτον, να διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόσβαση στις αγορές για κάποια προϊόντα από την Ουκρανία, εφόσον βέβαια πληρούν τα πρότυπά σας. Και τέλος, να απελευθερωθεί πολύ πιο γρήγορα η μακροοικονομική βοήθεια προς την χώρα μου και να ε, αρχίσουν να λειτουργούν και πάλι τα προγράμματα ε, η βοήθεια στον προπολογισμό. Ελπίζω να δείξει θάρρος αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου χώρα θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όπως είχε συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών του 2012. Ακόμα και χθες έγιναν υψηλού επίπεδου διαβουλεύσεις ε, στις Βρυξέλλες που ε, είπαν ότι βρισκόμαστε στην καλή πορεία. Φίλοι μου, 22 χρόνια γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την εξαρτησία μας και ο πρόεδρος είπε σαφώς. Για την Ουκρανία η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μία μια μεγάλη κινητήρια δύναμη για να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πιο ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος. Λοιπόν, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Να το προσέξουμε, προσέξτε το παρακαλώ και σας ευχαριστώ κύριε Πρόκ που αυτή την έγκυρη συζήτηση τη διοργανώσατε. Thank uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για την κρίση ανάμεσα στην Ουκρανία ε, και την Ρωσία, σε εμπορικές του σχέσεις δηλαδή, που εξεράγει τον Αύγουστο. Δυστυχώς αυτό συνιστά παράδοση ε, ε, είτε τον Αύγουστο είτε το Δεκέμβρη ανακύπτουν τα σοβαρά ζητήματα. the e ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την ιστορία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δεκάδες συμφωνίες ε, σύνδεσης και ελευθέρων εμπορικών ε, συναλλαγών. Πρώτη φορά όμως έχουμε τέτοια αντίδραση τρίτου μέρους κατά μιας τέτοια συμφωνίας. Εξυπακούεται ότι δεν πρόκειται για νέα και να πάντα είχε εξέλιξη. Από το 2007 έως το 2012 διήρκησαν οι διαπραγματεύσεις και αρχικά είχε προβλεφθεί για το 2012 υπογραφή της συμφωνίας ελπιστούμε τώρα ότι εντός ολίγων μηνών θα ε, προσπογραφεί. Και βλέπουμε λοιπόν μια ισχυρότατη αντίδραση κατά της βούλησης του Ουκρανικού λαού που ξεκίνησε αυτές τις διαπραγματεύσεις και εξάλλου οι διαδοχικές κυβερνήσεις της Ουκρανίας ε, ε, μετήχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο πρέσβης μας περιέγραψε την κατάσταση στα σύνορα με την Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, ε, εξομαλύνθηκε η κατάσταση από ό,τι φαίνεται ε, και η διακίνηση των προϊόντων είναι απαραίτητη για την οικονομία και των δύο χωρών και ελπίζουμε να παραμείνουν έτσι τα πράγματα εφεξής Τώρα, ως προς την αρχή, μία διμερή σχέση θα πρέπει να εξευρεθεί δυνάμει των υποχρεώσεων που έχουν αναλυφθεί ε, από αμφότερες τις πλευρές στα πλαίσια του ΠΟΕΜ διότι ε, οι εμπορικές του σχέσεις διέπονται από τους κανόνες ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπόριου. Τώρα οι εξελίξεις τις τελευταίες ε, δύο εβδομάδες δυστυχώς έδειξαν ότι ε, είναι ε, αδιαμφισβήτη η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ανοιχτά ασκεί πίεση η Ρωσία επί της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο υπογραφής αυτής της συμφωνίας σύνδεσης όπου συμπεριλαμβάνεται και αυτή η σφαιρική και σε βάθος Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών από το Κρεμλίνο επίσημες πηγές ε, κοινοποίησαν ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ε, θα ενεργοποιηθεί μία ε, μόνιμη εντατικοποίηση, αν θέλετε, των τελωνιακών ελέγχων. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα ήταν ε, αυτοκτονία για την Ουκρανία να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εάν υπογράψει δε τη συμφωνία το Κίεβο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να μετάσχει στην Τελωνιακή Ένωση, της οποίας ηγείται η Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, στη Μόσχα τη Δευτέρα προσθέθηκε ότι θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα για την Ουκρανία και η Ρωσία, πάση θυσία, θέλει να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο. τέλο παράθεσο. Ο ίδιο ο πρόεδρος Πούτιν την περασμένη εβδομάδα ε, ξέφρασε την άποψή του ότι η Ρωσία θα αναλάβει προστατευτικά μέτρα για να προστατεύσει τις αγορές της ε, λόγω των όρων που θα επικρατήσουν εάν υπογραφεί η συμφωνία. Δεν υπάρχει συνοριακή διένεξη ε, επίσημα, αλλά σίγουρα θα αρχίσει μία διαδικασία που δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πλήρη διαβούλευση με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα διαστόματος του εμπορικού της αντιπροσώπου και χθες ε, διαστόματος του Επιτρόπου Φίλε. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις στο ζήτημα. Είναι κυρίαρχη η χώρα η Ουκρανία και άρα μπορεί να κάνει ελεύθερα τις επιλογές της ως προς τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Ε, παρέ Έγινε παραπομπή επίσης ε, στην ε, τελική πράξη της συμφωνίας ε, του Ελσίνκη που είναι και η βάση στην οποία εδράζεται η συνεργασία και η σύνδεση όχι μόνο με την Ουκρανία αλλά και με την Ρωσική Ομοσπονδία. Επανειλημμένα οι Ουκρανοί επανέλαβαν τη βούληση τους να ακολουθήσουν αυτήν την ρότα της υπογραφής συμφωνίας σύνδεσης διότι αυτό συνιστά, έχει ρόλο κλειδί μάλλον για τον εκδημοκρατισμό για και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Σε καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν παρεμποδίζει την Ουκρανία από το να ε, αναπτύξει μια επικοδομητική σχέση με την Τελωνιακή Ένωση στην οποία μετέχει η Ρωσική Ομοσπονδία στο μέτρο που γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του ΠΟΕ και στο μέτρο που δεν παραβιάζεται η σφαιρική και εις βάθους ε, ε, συμφωνία ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών. Τώρα, οι εμπορικές απειλές από πλευράς της Ρωσίας ε, που ασκούνται ε, για να αποτραπεί η υπογραφή είναι μια παράδεκτη εξέλιξη και τονίζουμε ότι η Συμφωνία Σύνδεσης ε, θα υπογραφεί επί τη βάση της απτής πρόοδου που έχει ε, σημειώσει η Ουκρανία και που διαπιστώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και θα επιβεβαιωθεί ελπίζουμε στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Ε, αυτά τα ορόσημα και ε, που χρησιμοποιήθηκαν για να κρυθεί αυτό δεν επηρεάζονται από τις τελευταίες εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρές εμπορικές ανησυχίες εξάλλου στις σχέσεις και με τη Ρωσία αλλά και με την Ουκρανία και ευελπιστεί ότι σύντομα θα εξευρεθεί μία λύση ούτω ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερότητα τη Ρωσία και τη Ουκρανία και η συμμόρφωση με τι ε, δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ουκρανία κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Επίση, ο σύμβουλο για θέματα εθνική ασφάλεια του Πρέδρου τη Ουκρανία, ο Άντρεϊ Κλούγεφ και ο υπουργό Δικαιοσύνη συναντήθηκαν με ε, ανώτατου εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέτασαν διεξοδικά ε, τα κριτήρια αυτά, ξεκάθαρα υπήρχε ένα μήνυμα υποστήριξη για τα εμπορικά ζητήματα και τα προβλήματα που ανέκυψαν πρόσφατα. Όμω ε, ε, υπήρξε και υποστήριξη για τις ε, προϊούσες ε, δυσκολίες εμπορικού χαρακτήρα που πρέπει να ρυθμίσουμε σε σχέση με την Ουκρανία για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι προς συμφέρον της Ουκρανίας να αναλάβει συγκεκριμένη δράση ούτως ώστε να ε, απόσχει από την ανάληψη προστατευτικών εμπορικών μέτρων αυτά κυρίως σε σχέση με το κόκο, τον άνθρακα και τα αυτοκίνητα. Επίση, υπάρχει το θέμα τη ευθυγράμμιση των δασμών μετά την προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορία. Έχουν αυξηθεί οι δασμοί σε πολλούς τομείς έκτοτε. Ε, τώρα αυτέ τα, διμερεί προβλήματα με την Ουκρανία έχουμε τη διευκόλυνση τη διακίνηση ουκρανικών προϊόντων. Αυτό είναι δυνατόν και ισχύει ήδη για κάποια ευαίσθητα προϊόντα. Αυτό εφάνει εξάλλου διότι η Ουκρανία είναι στον ε, κατάλογο των χωρών που μπορούν να εξάγουν πουλερικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση τώρα με τη Ρωσία και την απόπειρα να περιορίσει τις εξαγωγές της ε, Ουκρανίας ε, σε σχέση με γνώμονα την ποιότητα ή την ασφάλεια είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε σε σχέση με τους κανόνες προέλευσης γιατί ακούστηκε και το επιχείρημα ότι ε, ξαφνικά θα πλημμυρίσει η ρωσική αγορά με προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Τουρκίας. Ε, κοιτάξτε, αυτή η ζώνη, ζώνη ελευθέρων συναλλαγών καλύπτει ούτως ή άλλως εξαγωγές, τις μελλοντικές εξαγωγές ε, της Ουκρανίας. Δεν θα υπάρχει όμως προτιμησιακό καθεστώς όταν οι εξαγωγές είναι προς την Ρωσία. Ξαναλέω, δεν θα υπάρχει προτιμησιακό καθεστώς για τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, διότι δεν προέρχονται προϊόντα από την Ουκρανία, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τελωνιακή της Ένωση. Ω εκ τούτου, με την υπογραφή τη συμφωνία με ένα τρίτο μέρο του τέστην με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ω ε, πρόσχημα, ούτε και η Ρωσία, για να εντατικοποιηθούν οι τελωνιακοί έλεγχοι. Τώρα, οι τελωνιακοί έλεγχοι ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσική Ομοσπονδία αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, που δραστηριοποιούνται και στι δύο αυτέ χώρε. Ε, επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε αυτές τις χώρες ε, και που έχουν ε, πολύ εξειδικευμένες συνιστώσεις για την παραγωγή τους επί το που Θέλουμε πάση να αποφύγουμε εμπορικό πόλεμο με τους δύο εταίρους μας. Έτσι θα πρέπει να διεκπαιρώσουμε αυτά τα ζητήματα εφαρμόζοντας τα πρότυπα του ΠΟΕ. Θα ήθελα δεν να τονίσω πως ε, η συμφωνία σύνδεσης ε, ε, δεν θα είναι εις βάρος των διμερών σχέσεων της Ουκρανίας με Ρωσία ή με άλλες γειτονικές χώρες. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι προσφέρει πολλά ωφέλη και πολλές νέες ευκαιρίες για την Ουκρανία και τους οικονομικούς τους φορείς, είτε είναι Ρώσοι, Τούρκοι, Ευρωπαίοι ή οποιασδήποτε άλλης υπηκότητας. Να υπογραμμίσω εν τέλει ότι θα παρακολουθούμε εκ του την κατάσταση και ε, στο ενδεδειγμένο επίπεδο θα συνεχιστεί ο πολιτικός ε, διάλογος με όλους εμπλεκόμενους φορείς. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο για όλες τις εξελίξεις και συγκεκριμένα και την, αρμόδια, την καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή ε, Εξωτερικού Εμπορίου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα υπολείπεται λίγοστό χρόνος. Ε, και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι πολύ σύντομες ε, οι παρεμβάσεις. Ε, θέλω να κλείσει τώρα ο κατάλογος των ομιλητών. Δέκα ομιλητές έχουμε. Και ο τελευταίος είναι ο Ντένις από τους Πρασίνους. Έκλεισε ο κατάλογος. 1,5 λεπτό και μετά θα περικόψουμε αν δεν προλαβαίνουμε. 1,5 λεπτό. Σάρις Βόλσκι. Θα εκφραστώ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ ε, τον Πρόεδρο που επέτρεψε να γίνει αυτή τόσο επίγουσα συζήτηση. Χαίρομαι που ήταν δυνατό να ε, εκφραστούμε από αυτού. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπροκ και τον κύριο Σβόμποντα, τον πρόεδρο των Σελδημοκρατών. Ξέρουμε ότι τον Αύγουστο πάντα προκύπτουν εκπλήξεις. Η Ρωσία ε, αρέσκεται πολύ σε τέτοιες αυγουστιάτικες εκπλήξεις. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα εμπορίου. Στην ουσία δεν πρόκειται καθόλου για θέμα εμπορίου. Πρόκειται για την ε, συνολική εταιρική σχέση μας προς Ανατολάς ε, για την Ουκρανία, δηλαδή την Αρμενία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των μέτρων αυτών, ε, θα υπάρξει και συνέχεια. Είναι γεωπολιτική λοιπόν η φύση της πρόκλησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σε πορεία σύγκρουσης. Χρησιμοποιείται η ήπια ισχύς για να επηρεαστεί η κατάσταση στην περιοχή. Πάντα υπάρχει αυτή η διάσταση στις σχέσεις ε, Ρωσίας-Ουκρανίας στο φυσικό αέριο. Και να μην ξεχνάμε ότι στην Μολδαβία υπάρχει η σύγκρουση στην Τρανσνιστρία. Ε, και είναι ένα μήνυμα και προς την Αρμενία αυτό. Βεβαίως να μην, ε, ε, μπορεί να μην υπάρχει εμπάργο, αλλά οι επιπτώσεις του εξακολουθούν. Και ε, και οι δύο πλευρές είναι πολύ πιθανό να λάβουν μέτρα. Αν υπάρξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ένωσης Ουκρανίας. Είμαστε λοιπόν εμπλεκόμενοι, δεν μπορούμε να είμαστε μόνο παρατηρητές. Και η Ένωση και η Ουκρανία έχουν δικαίωμα επιλογής των εμπορικών τους εταίρων. Η Κομισιόν πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά την κατάσταση, να μην αντιμετωπίσει το θέμα αυτό ως καθαρά εμπορικό θέμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πίεση των Ρώσων, η Ουκρανία έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές της ελεύθερα και γι' αυτό θα πρέπει να ξανατονίσουμε τις τρεις απαιτήσεις στην Ένωση. Η κυρία Τιμοσέγκο πρέπει να απελευθερωθεί, να υπάρξει μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού συστήματος και η Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερες διπλωματικές ενέργειες έναντι της ε, Ρωσίας. Και στα πλαίσια του G20 πρέπει το θέμα να συζητηθεί. Στην Ολομέλεια να υπάρξει ψήσμα, γι' αυτό προτείνω, για το θέμα πιέσει από τρίτες χώρες σε περιπτώσεις συμφωνίων, συμφωνιών Γεια σας. Το Γιάτσικ μάλλον δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Ελπίζω οι επόμενοι ομιλητές, ε, ε, να, οι επόμενοι ομιλητές να σεβαστούν περισσότερο τις ε, προϋποθέσεις που έχω θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ε, διαφορές απόψεων μεταξύ ημών για το θέμα αυτό. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και ο κύριο Βόλσκι περιγράφουν ε, σαφώς και ακριβώς τους μηχανισμούς ε, που έχουν τεθεί εν Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν στόχο το Κρεμλίνο να ε, επηρεάζει τις αποφάσεις για τα οικονομικά θέματα των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Όσο δεν υπήρχε κίνδυνος ε, να λάβει τέτοιες αποφάσεις η Ουκρανία, ε, τόσο περισσότερο ε, βασίζεται σε εκδηλώσεις ήπιας ισχύω. Όμως υπάρχει μια εκστρατεία χρηματοδοτούμενη με ρωσικό χρήμα που προσπαθεί να πείσει την Ουκρανία ότι δεν πρέπει και τον πληθυσμό της Ουκρανίας ότι δεν έχει και πολλά να περιμένει από περισσότερες σχέσεις με την Ένωση. Τώρα όμως εντελώς ξεδιάνθρωπα και ανοιχτά προσπαθεί η ρωσική πλευρά μέσω ε, δραστικών μέτρων ε, που ε, δημιουργούν τεράστιες δυσχέρειες στην Ουκρανία και δεν αφορά μόνο την Ουκρανία και την κυβέρνηση αφορούν ακόμη και επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και άλλες επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς πολίτες που διαπιστώνουν ότι το μέλλον τους είναι σε κίνδυνο. εφόσον θέλουμε ε, να θεωρούμεθα ε, πολιτισμένες χώρες, πρέπει να εγγυόμεθα όχι μόνο τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές ελευθερίες. Πρέπει οπωσδήποτε η Ουκρανία να τηρήσει αυτούς τους κανόνες. Ευχαριστώ κάπως καλύτερα τα πήγαμε από πλευράς χρόνου, λέει ο Πρόεδρος. Η Ρεμπέκα Χάρμς οπωσδήποτε θα θα κάνει, τα πάει ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ε, πρόκληση λόγω αυτών των εξελίξεων που δημιουργούν τέτοια έκπληξη. Η ομάδα μου όμως ε, δεν τα θεωρεί και τόσο αναπάντεχα αυτά που κάνει τώρα η Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα σε αυτή τη σύγκρουση με περίσκεψη. Θέλουμε η Συμφωνία Σύνδεσης να βοηθήσει ε, να υπάρξει στην Ουκρανία οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη δημοκρατία. Αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης ποτέ δεν θεωρήθηκε από πλευρά μα ω όπλο κατά τη Ρωσία. Σε πολλέ συζητήσει ε, είπα στου Ουκρανού και στο Κίεβο ότι είμαι πεισμένη ότι Και τους είπα λοιπόν ότι όπως και εμείς ε, ως Ένωση χρειαζόμαστε οικονομικές σχέσεις με την ε, Ρωσία, τόσο τις χρειάζεται και η Ουκρανία. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτή η σύγκρουση με τη Ρωσία πρέπει να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς, είναι απαράδεκτο, είναι καθαρή παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ, όμως δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουμε με τις απαιτήσει μας για τις σχέσεις μας με την Ουκρανία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Ρωσία. Το πρόβλημα είναι ε, ότι οι απαιτήσει μα για την απελευθέρωση τη κυρία Τιμοσέγκο για μεταρρύθμιση του νομοθετικού συστήματο είναι προποθέσει. Πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθούν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά στο Βίλνιους για την Ευρώπη και την Ουκρανία. Ο κύριος Κόμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως έχουμε να κάνουμε εδώ όχι μόνο για την Ρόσελ και άλλους μεγάλους Ουκρανικούς ομίλους. Μιλάμε και για θέσεις εργασίας για τους Ουκρανούς. Μιλάμε όμως και για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας. Τι κάνουμε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που τώρα βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία και ζητούμε από την Ουκρανία να κάνει τελευταία που αρμόζει να κάνει, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαστικό σύστημα και μήπω θα μπορούσε να πει κανένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα θα ήταν να μην έχει τη συμφωνία με την Ουκρανία. Η απάντηση όμω είναι απλή. Χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία. Είναι υπέρ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για μα θα υπάρχουν θετικά σημεία από αυτή τη συμφωνία. Είναι λοιπόν σαφή η κυρία μα θέση και έτσι θα τα πούμε ε, προς το Κίεβο. Από τη μια βέβαια θα επικρίνουμε τη Ρωσία, από την όλη όμω θα δούμε και εμεί τι μπορούμε να κάνουμε. Και ε, από αυτό που θα γίνει τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι. Ίσως θα σοκάρω κυρίες και κύριοι ότι θα πούμε ότι δεν θα πρέπει στη Βίλνα να αφήσουμε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Αύριο μεθαύριο θα πρέπει να υπογραφεί στο Κύβο και στις Βρυξέλλες, να γίνει αυτό το σωμότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση γύρω από τη συμφωνία. Θα πρέπει να επιληθούν τα θέματα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και τη Ρωσία και από την άλλη και η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουν να συμμορφωθεί η Μόσχα. Ε, κύριε Λίσεκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Ουκρανό πρέσβη που τόνισε τις επιλογές της χώρας του. Να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέφερε ότι δέχεται η χώρα, δέχεται Ουκρανία πιέσης από τη Ρωσία. Να σας πω όμως από την άλλη με με αυτά που είπε ο πρόεδρος Πούτιν. Να, γιατί να μην τον προτείνουμε να, για το Νομπέλ ιατρικής, ιδιαίτερα για το τομέα της οφθαλμολογίας. Γιατί άνοιξε τα μάτια όλων μας που μέχρι τώρα δεν έβλεπαν ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο ε, της Ρωσίας. Τώρα πλέον σε όλη την Ευρώπη είδαμε το φως το αληθινό, είδαμε το στόχο της Ρωσίας. ναι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μέσα εισαγωγές, εισαγωγές ε, χάλιβα και φυσικού αερίου. Από την όλη όμως μην ξεχνάμε τη ζωρική αυτή τη στιγμή για την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, πόρτα για την Ουκρανία. Ο κύριος Σιλεύκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ να κάνουμε με μια σοβαρή προσπάθεια να περιοριστεί η εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας. Αυτή η κρίση όμως δεν αφιβόλω και την εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μετέχει στην όλη υπόθεση Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε μόνο ότι είναι καθαρά θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αντιδράσει στεναρά. Και το Ευρωκοινοβούλιο μάλιστα θα πρέπει στεναρά να αντιδράσει. Χρειαζόμαστε πιστεύω εγώ μία απόφαση αυτό να το προετοιμάσουμε για το Στρασβούργο όπου να, με ένα ψήφισμα να καταδικάσουμε την προσπάθεια ανάμειξης της Ρωσίας και να πούμε σαφέστατα ότι το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να ξεκινήσει πιο πρώιμα προσωρινά ή συμφωνία για την ελεύθερη ζώνη συναλλαγών. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει να λειτουργεί η συμφωνία σύνδεσης και θα πρέπει να αφήσουμε καμία αμφιβολία σχετικά με τη θέση μας ότι είμαστε υπέρ της συμφωνίας σύνδεσης και ότι θα πρέπει να υπογραφεί αυτό το φθινόπωρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Τρανσμπέργκης. Ευχαριστώ Έλμαρ. Εμείς, η Ευρώπη εννοώ, είμαστε σε πολύ ενώπιν μιας πολύ κρίσιμης υπόθεσης. Ένα σταυροδρόμι και για την Ουκρανία, αλλά μάλλον και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε πάντα να καθησυχάζουμε τα πράγματα με τα όσα κάνει η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία θέλει να προσπίσει όλα τα συμφέροντά της. Δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να προσπίσει τα συμφέροντά της όταν αυτό σημαίνει ότι περιορίζουν άλλων ελευθερίες. Θα πρέπει αυτές οι ελευθερίες να είναι κάτι που προσπιζόμαστε. θα πρέπει να είναι ελεύθερη να επιλέξει Ουκρανία. το τάδε υπογραφή ή όχι συμφωνία έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι δύο πλευρές που διαπραγματεύονται. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει συμφωνία εάν και η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδείξουν επαρκή θέληση για συνεργασία και να απορρίψουν οποιαδήποτε εξωτερική απειλεί η πίεση. Θα πρέπει αυτή τη θέληση όμως να τη δείξουμε. Να τη δείξουν και οι δύο πλευρές. Δεν μπορούμε να δείξουμε ότι δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Και στην Ουκρανία υπάρχουν ε, δυνάμεις που αντιδρούν. Φυσικά ε, της υποκίνει η Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι με θετικό τρόπο. Όλα θα πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Λέω κύριο κύριος Ε, πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο πως ε, δυσχερέδουν οι σχέσεις διαρκώς, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα με τη Δύση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι διμερείς σχέσεις Αμερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της υπόθεσης Νόντεν επιδεινώνονται ε, διαρκώς και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάσουμε επίση την κατάσταση στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εισερχόμεθα σε μια περίοδο ε, έντασης, ε, κρίσης, όπως το 2009. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν αυτό ισχύει. Ευχαριστούμε, Μπίλαν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται μια ταχύτατη αντίδραση. Και εσείς το κάνατε αυτό, ταχύτατα ε, συγκαλέσατε αυτήν την συζήτηση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι προφανές ότι οι συγκρούσεις αυτές ε, πολύ συχνά ξεκινάνε από τη Ρωσία. Ε, και μάλιστα γίνονται τον Αύγουστο, όταν εμείς είμαστε σε διακοπές. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Ευχαριστώ λοιπόν τον Έλμαρ Μπρουκ που επέτρεψε να γίνει αυτή η συνεδρίαση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της θέσης της. Είναι προφανής λοιπόν έλεγα η προθέση της Ρωσίας ένας από τους συμβούλους του Πρόεδρου Πούτιν, Σεργέη Αγκλάζιεφ, είπε σαφώς πρόκειται για προσπάθεια εκβιασμού. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει εμφιβολία ότι δεν είναι θέμα μόνο εμπορικών σχέσεων. Η Ρωσία αξιοποιεί όλα τα παραδοσιακά μέσα, ανεβαίνει τιμή του φυσικού αερίου, αλλά εδώ ε, ε, ασκούνται και ευρύτερε γεωπολιτικές πιέσεις για ευρύτερους τέτοιους λόγους. Ε, οπωσδήποτε εμπλεκόμεθα σε αυτήν την ε, ε, σύγκρουση γιατί υπάρχει συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Γι' αυτό η αντίδραση της Ένωσης πρέπει να είναι αποφασιστική και σαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή μας και βεβαίως και η Ολομέλεια πρέπει να καταστήσουν σαφή τη θέση μας και μια ερώτηση προς τον Ουκρανό πρέσβη. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του, για τις παρατηρήσεις του. Χαιρετίζουμε το ότι είναι αποφασισμένη να υπογράψει αυτή τη συμφωνία η Ουκρανία, αλλά ε, ε λαμβάνουμε και ορισμένα μηνύματα που μπορούν να παρερμηνευθούν από τους αντιπάλους της Ουκρανίας. Ο κύριος Αζάροφ, για παράδειγμα, είπε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να συνάψει και άλλες συμφωνίες. Τι σημαίνει αυτό. Η κυρία Όμιν θα είμαι σύντομη έχουμε να κάνουμε μια εμπορική σύγκρουση αυτή τη στιγμή, η οποία καταρχήν θα μπορούσε να επιληθεί στα πλαίσια του Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Εμπορίου. Μετά θα υπάρχουν συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να επιλύσουμε τα πράγματα βέβαια γιατί θέλουμε να περάσει από το Κοινοβούλιο το θέμα της, πολιτικ... της ε, Νοέμβριο. Αυτές θα, έχουν και, θα έχουμε και πολιτικές όμως συνέπειες για εσάς, ε, διότι ακόμα χωλαίνει το κράτος ε, δικαίου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η εμπορική σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να επιλύσετε τα θέματα σε αυτό το σημείο του χαρτοπορίας, το άλλο που ανέφερε η Ρεμπέκα να αναλάβετε νέες δράσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. The last one, Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντένις Μέκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω να υπάρχει μεγάλη σύμπνια και αυτό με ικανοποιεί. Εγώ είμαι υπέρ τη άποψη ότι φυσικά θα πρέπει να είναι πλήρως ελεύθερη να αποφασίσει για το τι κάνει η Ουκρανία ανεξάρτητε αποφάσει να παίρνει. Είναι απαράδεκτο που αναμειγνύεται η Ρωσία. Πολύ συχνά πήγα τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία και αυτό το καλοκαίρι πήγα όταν ε, είχε γίνει αυτός ο μίνι εμπορικό ε, πόλεμο. Ε, είναι αυτό μια έκφανση μια ανοιχτή πλέον στρατηγικής της Ρωσίας, γεωστρατηγικής, δεν το κρύβουνε άλλωστε. Διάβασα χθε ε, στο, στο ρωσικό ε, ένα ρωσικό περιοδικό, το Second Daily, ένα άρθρο που έλεγε καθαρά ποια είναι η στρατηγική του. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, έχει πολλές δυνατότητες, έχει έναν φιλόπονο πληθυσμό, έχει ανάγκη αυτή η χώρα και επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που κάνει η Ρωσία δεν είναι, δεν είναι πολιτική καλής γειτονίας. Είναι και τα διασωρικά προβλήματα βέβαια που έχει ανέκαθεν η Ουκρανία με την Ρωσία. Μην ξεχνάνε όμως οι Ρώσοι ότι πάντα θα παραμείνουν γείτονες ε, της Ουκρανίας να αποφασίσουν αν θα είναι καλοί γείτονες ή κακοί γείτονες. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα εντυπωσιάζομαι από την πλήρη υποστήριξη από πλευρές του Κοινοβουλίου για την θέση της Ουκρανίας, για την υπογραφή πρώτα απ' όλα της συμφωνίας ε, ε, σύνδεσης Καθώ και σε σχέση με την διένεξη με τη Ρωσική Ομοσπονδία για τα εμπορικά και τελωνιακά ζητήματα. Καλωσορίζουμε την ε, απερίφραστη υποστήριξή σα. Δεύτερον, παρακαλώ να λάβετε υπόψη τις συστάσει στι οποίε αναφέρθηκα στην πρώτη μου παρέμβαση, αυτά τα 7 σημεία που ανέφερα παρακαλούμε να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο και από την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Τρίτον, θα ήθελα να σας καθησυχάσω και πάλι σε σχέση με την δέσμευση της Ουκρανίας ε, για ε, απτή πρόοδο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα συγκεκριμένα κριτήρια του συμπεράσματος του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2012. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, διαφωνία με την Ρωσία για να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το Δεκέμβριο του 2012. Είναι ισχυρή η δέσμευσή μας και έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω ε, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή σας ε, για την υποστήριξή σας. Μπορείτε να υπολογίσετε σε εμά. Ε, με οικοδομητικό πνεύμα συνεχίζουμε την συνεργασία και τις διαβουλεύσεις με τη Ρωσία για να διεκπαιρεώσουμε αυτά τα εκρεμή ζητήματα στα πλαίσια της ε, εταιρική στρατηγικού χαρακτήρα σχέσης μας. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Είναι ευρία η συνάντηση εδώ διαπιστώνω ως προς την πολιτική σημασία των πεπραγμένων ε, και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούμε την υπόθεση. Οι δεσμεύσει ε, στου κόλπου του ΠΟΕ θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και φυσικά βάση της τελικής πράξης συμφωνίας του Ελσίνκη θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της ελεύθερης επιλογής ε, των χωρών. Ε, αυτές οι αρχές θα πρέπει να μας καθοδηγούν. Δεν είναι προς κάθε ενός να δημιουργούμε τεχνητές ε, πολιτικές πιέσεις και οικονομικές δυσκολίες. Είναι προς συμφέρον όλων να είναι ελεύθερες οι επενδυτικές και εμπορικές ροές προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδιστούν σε καμία περίπτωση το αντίθετο να ενθαρρυνθούν σε όλα τα επίπεδα θα ε, ε, συνεχιστεί η συζήτηση και ελπίζω και ε, στην συνεδρίαση G20 να ασχοληθούν έστω και ακροφυγώς με αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους όλους. Όπως βλέπετε υπάρχει ευρεία συνένεση. ότι πρώτον ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να δρά όπως δρά και δεύτερον θέλουμε να υπογραφεί στο Βίλνιους η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία. Τρίτον ελπίζουμε η κυβέρνηση της Ουκρανίας να έχει τη δυνατότητα να την υπογράψει. Αυτά είναι τα τρία σημεία επί των οποίων συμφωνούμε και υπάρχει οπωσδήποτε και ελπίδα αλλά είναι αναγκαίο να γίνουν αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους συναδέλφους ε, Γιασένιου και Κλίτσκο ε, να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε προβλέψει μισή ώρα για το θέμα αυτό. Να υπάρξει μια παρουσίαση εισαγωγική 10 λεπτών και μετά να υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Διότι πρέπει 12.30 να τελειώσουμε ακριβώς. Βιτάλη. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Πολύ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία σήμερα να λάβω μέρος συνεδρίας σας, να σας μιλήσω. Το κόμμα μας είναι πολύ ικανοποιημένο για την προσοχή που δίνει στα θέματα της Ουκρανίας διαρκώς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο σήμερα είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι πιο πρόσφατες εμπορικέ κυρώσεις της Ρωσίας κατά της εκκρονίας που παραβιάζουν πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες όπως και τους κανόνες ε, του ε, ΠΟΕ. Δεν είναι να μπορεί κανένας από όσο ξοργίστηκαν οι Ουκρανοί κατά αυτών των δράσεων. Καταδικάζουμε σαφώς ε, την κατάσταση και τις πράξεις της Ρωσίας. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια πράγματα οι ρωσικές αρχές. Αλλά μέχρι τώρα δεν το είχαν κάνει τόσο κοινικά και τόσο συστηματικά ταυτόχρονα. Προσπαθούν να απειλήσουν την Ουκρανία, να υποσκάψουν την συμφωνία δέσμευσης, να εμποδίσουν την δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερης συναλλαγών. Και ούτε καν πλέον κρύβει η ρωσική κυβέρνηση στους γεωπολιτικούς ε, στόχους. Στην επόμενη κοινή μας συνεδρία θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και Νομίζουμε ότι θα πρέπει όλα τα μέσα να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία για να προσφύγει τα συμφέροντά της απέναντι ε, στην Ρωσία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προασπιστεί τις πολιτισμένες αρχές της σχέσης ανάμεσα σε χώρες. Ε, αυτές οι εμπορικές κυρώσεις που επιβάλλει η Ρωσία δείχνει βέβαια το πόσο μεγάλη σημασία έχει υπογραφή της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης. Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτή της συμφωνίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην εξέλιξη της χώρας μου αλλά θα έχει επιπτώσεις και σε πολλές άλλες χώρες ε, στην περιοχή. Βεβαίως εμείς είμαστε ρεαλιστές και καταλαβαίνουμε πλήρως ότι η επίτευξη του κοινού μας στόχου δηλαδή της υπογραφής της ε, συμφωνίας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμφωνία ε, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς να εκπληρώσουμε τους όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φελεύουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει όλα τα βήματα που θα έπρεπε να είχε κάνει. Σε αυτό συμφωνεί όλη η πολίτευση και αυτό θα το επαναλάβουμε και πάλι στην επόμενα συνεδρίαση ότι θα πρέπει να ψηφιστούν οι απαραίτητοι νόμοι για την ε, ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας Ουκρανίας. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούν αυτά τα νομοθετήματα την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας πριν λάβει την οριστική απόφαση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο εργαλείο η μελλοντική συμφωνία για τον έλεγχο και την επιρροή στις δραστηριότητες της τωρινής Ουκρανικής κυβέρνησης. Θα ενισχύσει την προστασία των δημοκρατικών αρχών και θα μας δώσει νέες δυνατότητες το 2015 να έχουμε νέες δίκες εκλογές και στην περίπτωση ε, νίκη των ε, ε, των υποψηφίων που είναι υπέρ της μεταρρυθμίσεως αυτό θα βοηθήσει πολύ να διαμορφωθεί και το εκλογικό του πρόγραμμα. Από την άλλη, μία αποτυχία της Συμφωνίας Σύνδεσης θα ήταν εργαλείο στα χέρια της αυτακυρικής κυβέρνησης για να απομακρυνθεί όλο και περισσότερο από δημοκρατικές αρχές. Να σας διαβεβαιώσω ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση θα κάνει ό,τι μπορεί για να πιέσει την ε, κυβέρνηση να υπογράψει τη συμφωνία όπως πρέπει. διότι μας πεπισμένοι για το πόσο μεγάλη σημασία έχει. Ότι θα βοηθήσει και στο θέμα της ελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων στην Ουκρανία. Ιδιαίτερα την απελευθέρωση της Γιούλια Τιμοσέγκο. Αυτό είναι κύριο μέλημα των πολιτικών προτεραιοτήτων μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αρζένη Γιαυτσένιουκ. Είναι πρόεδρος της Μπατκιουσίνα, που είναι κόμμα... Είναι στην αντιπολίτευση, είναι το κόμμα της κυρίας Τιμοσέγκο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε ενώπιόν σας. Ε, θα ήθελα να είμαι σύντομος και περιεκτικός. Έχουμε αναλάβει σαφέστατη δέσμευση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πιστεύουμε ότι θα υπογραφεί η συνθήκη τον Νοέμβριο. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να τελεσφορήσει η προσπάθεια. Έχουμε ήδη καταθέσει μία σειρά από νομοσχέδια και ζητήσει από τον Πρόεδρο και τη Βουλή να εγκριθούν τα νομοσχέδια με τρόπο ώστε να συμμορφωθούμε βασικά κριτήρια που συνιστούν και ε, προϋποθέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας. Τρία κριτήρια και προϋποθέσεις σχετίζονται με δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανική κυβέρνηση πιστεύουμε θα εκτελέσει αυτά τα αιτήματα. Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι να σταματήσει η επιλεκτική δικαιοσύνη και να αποφυλακιστεί η Γιούλια Τιμοσέγκο. Δεύτερον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευελπιστούμε ότι θα της επιτρέψει να αποχωρήσει από τη χώρα για να τύχει ε, περίθαλψη στη Γερμανία. Δεύτερη προϋπόθεση για την εισαγγελία. Ε, έχουμε ακόμη το κληροδότημα από την ε, πρώην Σοβιετική εισαγγελία και βάσει των συμπειρασμάτων της Επιτροπής της Βενετίας θα ε, προταθούν και άλλα νομοσχέδια τα οποία θα υποστηρίξουμε ώστε να επικρατήσει το κράτος δικαίου και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την εισαγγελία. Τρίτο και ε, πολύ βασικό ζήτημα, πυλώνας κάθε δημοκρατικού κράτους, η εκλογική διαδικασία. Το 2012 έγινε η τελευταία ε, εκλογική αναμέτρηση και υπάρχουν ε, πέντε κομιτείες όπου είναι αμφιλεγόμενα τα αποτελέσματα. Έχουμε αναλάβει δέσμευση για επαναλάβει, ε, επανάληψη γνώμη της εκλογικής ε, αναμέτρησης. Βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με την ε, Ουκρανία, λένε κάποιοι. Όχι, θα διαφωνήσουμε. Είναι η γεωπολιτική κίνηση της Ρωσίας και δεν κατευθύνεται μόνο κατά της ε, Ουκρανίας αποδέκτες είναι και η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από κοινού, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε μια κρατεά απάντηση. Οι βαλτικές χώρες, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έκανε η Ρωσία προτού προσχωρήσουν στην Ένωση και στο ΝΑΤΟ τι έγινε. Ε, στη, στο Βουκουρέστι το 2008 στη Σύνοδο η Ουκρανία ζήτησε σχέδιο δράσης για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Τότε το ίδιο έκαναν. Ανέλαβαν ε, παρεμφερείς δράσεις τότε και το κλειδί για μας είναι ότι δεν είναι μόνο ζήτημα επιβίωσης, θέλουμε να ενισχυθεί το Ουκρανικό κράτος και να ενισχυθεί ε, να ενισχυθεί η θέση μας ε, ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Ρωσική Ομοσπονδία παραβίασε μια σειρά από διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Έχουμε τους κανόνες του ΠΟΕ, Στη συνέχεια έχουμε τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία που εγκρίθηκε από τη Βουλή μας πριν από λίγους μήνες. Αλλά ξαναλέω το ζήτημα δεν είναι το εμπόριο, είναι η γεωπολιτική και ο πρόεδρο Πούτιν ήταν ξεκάθαρος. Θεωρεί ότι η Τελωνιακή Ένωση δεν είναι οικονομική. Είναι πολιτική ένωση. Εγώ θεωρώ ότι η Ρωσική Ομοσπονδία και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει μια νέα, ε, τη Σοβιετική Ένωση, μια νέα εκδοχή. 2-0. Εμείς 80 ε, χρόνια και βάλει ήμασταν σε αυτή την ένωση. Φτάνει. Τώρα θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η καλύτερη ελπίδα που έχουμε είναι να υπογραφεί και να εκτελεστεί αυτή η συμφωνία. Η Ουκρανία ελεύθερες ε, και δίκαιες ε, προεδρικές εκλογές χωρίς αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να έχει. Αυτό είναι άλλο ένα εχέγγυο για μας ε, πώς να είναι ελεύθερες και δίκαιες οι προεδρικές εκλογές που θα λάβουν χώρα στην Ουκρανία το 2015 η συμφωνία, η υπογραφή της συμφωνίας. Το μέλλον μας είναι ευρωπαϊκό. Είναι, έγκυται στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αναλάβει σαφή δέσμευση και θα ζητήσουμε επίσημα από την κυβέρνηση να ε, υλοποιήσει αυτά τα ε, τρία μέτρα στα οποία προαναφέρθηκα και θα προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας ε, για την επιτεύξη αυτού του στόχου. Θα επιτύχουμε ε, σε, αυτό το, σε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική που έχουμε ήδη θέση. Σας ευχαριστούμε κύριος ε, Σαρισβόλσκι. Χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει ενιαία άποψη της αντιπολίτευσης για αυτό, για το θέμα της ένταξης και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, για το θέμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, σύσφυξης των σχέσεων ακούγοντα ε, τους, ε, και τον πρέσβη προηγουμένως βλέπω ότι και αρχές είναι υπέρ αυτής της λύσης. Υπάρχει πρόταση από την αντιπολίτευση που μόλις είπε ο κ. Γιασένιουκ ότι στηρίζεται την κυβέρνηση σε όλες τις ενέργειές της για να εφαρμοστεί η συνθήκη ε, σύνδεσης και ακούστηκε και ότι για το θέμα αυτό η αντιπολίτευση ε, παρέχει περιορισμένη και υπό όρους εμπιστοσύνη ε, στήριξη στην κυβέρνηση. Χαίρομαι που έχει υπάρξει αυτή η ε, ομοφωνία για την σύσφυξη των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ένωση και χαίρομαι και για την εργασία που έχει κάνει το Κοινοβούλιο για να μεταγραφούν 1.200 νομοθετήματα της Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο. Έχουν αναφερθεί τα τρία κριτήρια, αλλά πριν το καλοκαίρι ε, υπήρξαν κάποια ανησυχητικά μηνύματα από τον Αράντα ε, ότι αναβλήθηκαν ορισμένα βασικά νομοθετικά βήματα. Χαίρομαι λοιπόν για τις δηλώσεις των κυρίων Κλίτσκου και Γιατσένιου ότι ε, θα επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι αν θέλουμε να επιτύχουμε το γενικότερο στόχο. Ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην πορεία σας ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη ε, όχι μόνο τι θα γίνει στι επόμενε εκλογέ, αλλά και τα συμφέροντα των επομένων γενεών. Η κυρία Μάιρεκ. Ο κύριο Μάιρεκ. Ευχαριστώ λοιπόν. Είναι συναρπαστικό να ακούμε τους κύριους Κλίτσκο και Γιατσένιουκ και συναρπαστικό να διαπιστώνουμε ότι είναι στο ίδιο ε, μήκο κύματο. Υπάρχει και άλλος αρχηγός της αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι παρόν εδώ. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και από τον τρίτο εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης για το ποια είναι η θέση του. Επί της ουσίας. Τις δηλώσεις αυτές τις θεωρώ ως σαφή ένδειξη από πλευράς ε, της αντιπολίτευσης και του ΕΛΚ, του οποίου είστε μέλη ή προσπαθείτε να γίνετε μέλη και θα ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αυτή για το θέμα συμφωνία σύνδεσης στην ε, ε, πολιτική σας ευρύτερη οικογένεια. Βεβαίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται θετικά η πορεία ε, σύσφυξη σχέσεων με την Ουκρανία αλλά βέβαια δεν είναι όλοι στον ίδιο βαθμό Ε, λίγο πριν την συνάντηση κορυφή στο Βίλνιου, γίνονται βέβαια ή μάλλον θα πρέπει να γίνουν ιδιαίτερες προσπάθειες από την πλευρά σας διότι η φωνή της αντιπολίτευσης είναι πολύ σημαντική για το θέμα αυτό. Το γεγονός ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος για το θέμα αυτό με την κυβέρνηση έχει μεγάλη σημασία. Το ότι υπάρχει ευρεία συνένεση. Και κάτι ακόμη. Είναι σημείο κλειδί αυτό για την ε, εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα θετικά ε, αλλά υπάρχουν και μερικά αρνητικά σημεία. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση ατόμων συγκεκριμένων, ε, συγκεκριμένου σεξουαλικού προσανατολισμού. Και θα ήθελα, εφόσον έχουμε εδώ μπροστά μας τους ε, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ίσως λοιπόν ε, θα ήθελα να τονίσω ότι ίσως θα έπρεπε να καλέσουμε και κάποιους από την ε, πλειοψηφία, το κόμμα των περιφερειών θα ήταν καλό για τα θέματα αυτά να ακούσουμε τις απόψεις όλων των πλευρών. Μα ήταν ο πρέσβη σήμερα παρόλο ο κύριος Μπροκ. Και ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Που εξεπροσώπησε την κυβέρνηση που ε, ε, στηρίζεται από, την, από το κόμμα των περιφερειών. Έχει ήδη έρθει εδώ λοιπόν εκπρόσωπος της κυβέρνησης και θα συνεχίσουμε να τους καλούμε και στους επόμενους δύο μήνες όταν θα πρέπει να πάρουμε απόφαση. Όσον αφορά το Βίλνιους και με ποιο τρόπο η κυβέρνηση ή το καθεστώς ε, στην Ουκρανία θα πιστούν να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις όπως το είπε και ο Σάιρος Βόλσκι, όπως το είπε και ο κύριος Βίγκαν, όπως και εγώ. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και με την σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Κράις Ντόφλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπορική πολιτική ανέκαθεν ήταν συνειφασμένη με την γεωπολιτική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στέγανα θέματα. Ε, αυτό το ξέρουμε από την εποχή της επικοκρατίας. Ε, Το θέμα είναι να υπογραφεί οπωσδήποτε αυτή η συμφωνία ε, αλλά θα πρέπει και οι δύο πλευρές να σεβαστούν του κανόνε. Δεν μπορούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επάνω κάτω τα καταθένα, τα, καταφέρατε ας υπογράψουμε στη Βίλνα. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο Πούτιν είναι να προβάλλει τα γεωπολιτικά του συμφέρονται. Και είναι σαφώς ότι δεν είναι αξιόπιστος εταίρο. Το θέμα είναι πώς γίνεται ο άλλος διάλογος. Τι λέει ο πολίτης στην Ουκρανία. Πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις κινήσεις της Ρωσίας. Γνωρίζουμε από την ιστορία, παραδείγματο χάρη, το φυσικό αέριο που έκοβαν στου ε, σκληρούς ε, χειμώνε. Πάντα άλλαζαν τις συμφωνίες που έχουν κάνει για να προωθήσουν τα δικά του συμφέροντα και φοβάμαι για το ότι ε, και όταν έχουμε τη συνάντηση στη Μόχα το G20 αναμένουμε με ενδιαφέρον το τι θα γίνει. Θα πρέπει και η ευρωπαϊκή πλευρά να δείξει ότι στηρίζει την Ουκρανία. Έχουμε αρκετές συγκρούσεις ε, και με τη Ρωσία ακόμα που του χρειαζόμαστε ως εταίρο. Αλλά όμως αναλάβει ανάλογη ευθύνη και ο Πούτιν. Και από την άλλη για τον ΠΟΕ παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι σαν να πνέει τα λίσθια θα έπρεπε κάτι να κάνει, να ξεκινήσει η διαδικασία παραβίασης κανόνων και στο πλαίσιο του ΠΟΕ. να μην πούμε ότι αφήνουμε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όταν υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης μετά όλα θα πάνε πολύ καλά. Ε, η κυρία Λουψέβα. Ελπίζω πάνω κάτω καλά να το είπα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, Σήμερα έγιναν ε, πολύ σοβαρές δηλώσεις και από την ε, Ουκρανική κυβέρνηση αλλά και από την Ουκρανική αντιπολίτευση. Διαπιστώσαμε λοιπόν σήμερα ότι και κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν στο θέμα την ίδια γνώμη. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς ε, για τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει όλα τα ενδιαφέρουνα μέρη να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χνοδιάγραμμα για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα πρέπει να υπογραφεί η Συμφωνία χωρίς όμως να πάρουμε κάποιες βεβαιωσμένες αποφάσεις. Έχω ε, μια ερώτηση για τους κύριους Κλίτσκο και για Τσένιουκ. Ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για από κοινού κινήσεις και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για να γίνουν σεβαστά τα κριτήρια και να υπογραφεί η συμφωνία. Μια άλλη ερώτηση. Ο πολίτης, η κοινωνία των πολιτών, τι άποψη έχει σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο κύριους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Καλό είναι που ακούμε ότι στηρίζετε πάντα την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας σας. είπα ότι ακόμα και αυτό το καλοκαίρι και πολλές φορές στο παρελθόν έχω πάει στην Ουκρανία και έχουμε τους πολίτες πολλές επαφές πάντα και ξέρω ότι στέκονται πίσω από την, στηρίζουν την ευρωπαϊκή πορεία. Έχω όμως και μια άλλη ερώτηση από την άλλη πλευρά, γιατί βλέπω να είναι επιφυλακτικοί οι πολίτες γενικώ απέναντι στην πολιτική, στους πολιτικοί στην Ουκρανία. Είτε μιλάμε για τους πολιτικούς της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης. Αρνητική στάση, μεγάλη επιφύλαξη, ε, καχύποπτη στάση και έχουμε μεγάλες βιβολίες για το πώς δημοκρατικές είναι εκλογές στη χώρα κατά πόσο γίνονται ελεύθερες εκλογές. Και αυτό βρίσκω ότι είναι επικίνδυνο όταν ο ίδιος ο πολίτης είναι καχύποπτος απέναντι στη δική του πολιτική τάξη. Αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Δεν ξέρω θα την επιβιώσετε εσείς ή όχι. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το πρόβλημα της διαφθοράς που από πάνω ως κάτω έχει διαποτίσει την κοινωνία και το σύστημα. Χρειάζονται, πιστεύω εγώ, μεταρρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη κασεκή νομοθεσία να είναι δίκαιη. Αυτό το θέλει πολύ ο πολίτης. Συμφωνείτε και εσείς και τι σκοπό έχετε να κάνετε. Ο κ. Μπέλο, κ. Προστακεύη, ζητήσατε με, αφού είχε κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών, τέλος πάντων. λιγότερο από ένα λεπτό αν είναι να σας δώσω τον λόγο για να απαντήσουν κιόλα οι προσκαλισμένοι. Κύριε Βίλαν, θα είμαι πολύ σύντομο. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία σε ό,τι αφορά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει δείξει ποια θα είναι τα τελικά της αποτελέσματα. Χαίρομαι που θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία αύριο ή μεθαύριο σε Βρυξέλλες και εκεί εγώ θα ήθελα εγώ να γίνει. Δεν θα γίνει όμως τόσο σύντομο. Μας μένουν δύο και περισσότεροι μήνες θρίλερ και πολέμου νεύρων, με αυτά που κάνει η Μόσχα, με την πολιτική που ασκεί όπως το βλέπουμε και τώρα. Χαίρομαι που σας άκουσα να λέτε πως η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση όπως το απορροσίασε ο κύριος Πρέσβης σε αυτό το θέμα μιλάνε με μία και μοναδική φωνή. Φυσικά θα πρέπει και οι κατάλληλε ομοθεσίε να περάσουν από τη βολή σα. Και η ερώτησή μου είναι ότι πραγματικά βρίσκεται και στην τελική ευθεία ό,τι αφορά στο να περάσουν αυτά τα νομοθετήματα από τη βολή και θα περάσουν τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση. Καλό είναι που είσαστε εσείς υπέρ ε, της υπογραφής των ζωμότερων δυνατών, όμως θα ήθελα να ξέρω και τη γνώμη σας σχετικά ε, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ασάροφ, αλλά και για το αν ε, θα συμμετάσχει η Ουκρανία σε διαφορετικές συμφωνίες στην ε, Τελωνική Ένωση με τη Ρωσία. Ε, αυτή τη στιγμή τι γραμμή έχει αυτό το θέμα η χώρα σας. 30 seconds, Mr. Κύριε Λαντσπέρκης, για 30 δευτερόλεπτα. Μα θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, θέλουμε, ε, επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ομοθυμία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπογραφή της συμφωνίας ε, και μεγαλύτερη ευελιξία για κάποιες ε, προϋποθέσεις. Θα δοθεί χάρη από τον τωρινό ή από τον μελλοντικό πρόεδρο στην Ιουλία Τιμοσέγκο κατά την αποφυλάκησή της και θα αποφυλακιστεί πριν ή μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι το σημαντικότερο σημείο. Εάν δεν υπογραφεί η συμφωνία στο Βίλνιους, αυτό είναι κακό και για την Ουκρανία και για τη Γιούλια Τιμοσέγκο. Και δεν θα έπρεπε να συμβεί. Thank you. Who starts now first? Σας ευχαριστούμε. Θέλετε πρώτο το λόγο. Ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο. You start now, this The other way around. So, uh, thank you for... Πολύ σημαντικές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Πρώτα απ' όλα, για τις μεταρρυθμίσεις ε, στην Ουκρανία. Για να είμαι ειλικρινή, το καλύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τη χώρα μου είναι να υπογράψουμε και να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης και την Σφαιρική και εις βάθος Συμφωνία Ελευθέρων ε, Εμπορικών Συναλλαγών. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό, έχει ήδη γίνει αυτό και το καλύτερο σχέδιο δράσης, ξαναλέω, είναι να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης και τη Σφαιρική Συμφωνία. Αυτό είναι πολύ πιο ευρωπαϊκό από οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να περάσουν 11 νομοσχέδια. Άρχισε μια στρογγυλή τράπεζα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη χώρα μου και όταν βλέπουμε ότι το Προεδρικό Επιτελείο, η Κυβέρνηση και η Επιτροπή των Περιφερειών ανήθηκαν να μετάσχουν σε αυτή τη στρογγυλή ε, τράπεζα, ε, θορυβηθήκαμε. Εκεί λοιπόν παρόλα αυτά θέσαμε ένα χρονοδιάγραμμα και καταθέσαμε σχέδια 11 νομοσχεδίων για να ολοκληρωθούν ε, οι δύο συμφωνίες ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης πλέον από πλευράς ε, του Προέδρου και της πλειοψηφίας Επιτροπής Περιφερειών. Προτίθενται να αναλάβουν πραγματικά ουσιαστικά βήματα και να περάσει νομοθεσία που πρέπει τόσο τον Οκτώβριο να υπογραφήσει συμφωνία. Τώρα για το ερώτημα για το πολιτικό βίο στην Ουκρανία και πώς εκλαμβάνει ο λαός ε, τις πολιτικές ε, φυσιογνωμίες. Ε, δεν μπορώ, εξαρτάται από τους πολιτικούς, δεν είναι να τους μισούμε όλους. χρειάζεται να κερδιθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια ευθύνη που βαραίνει τη νέα πολιτική τάξη της Ουκρανίας. Εμείς σε αυτό αποσκοπούμε και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δράσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη Συμφωνία Σύνδεση και τη Σφαιρική Συμφωνία για να δείξουμε στο λαό ότι είμαστε ε, φιλοευρωπαϊστές και να τους εξηγήσουμε με ποιου θα ε, συνεργαστούμε. Με εσάς, εσείς θα είστε οι εταίροι μας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επόμενο ερώτημα. Κοίταξε, είναι παράδοξο. Τελευταία δημοσκόπηση και όταν ο Γιανουκόβιτς ε, ανέλαβε την Προεδρία, έγινε επίση δημοσκόπηση και το 2009 και 2010, βάσει των δημοσκοπήσεων, η πλειοψηφία του Ουκρανικού λαού υποστηρίζει την ολοκλήρωση στην υπερεθνική ιονότητα που ελέγχει η Ρωσία. 56% ε, ο Γιαννουκόβιτς θεωρείται προ ε, ε, φύλλα προσκύμενου στους Ρώσους. 56% των Ουκρανών όμω σήμερα τετάχθησαν υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Λοιπόν, αυτά είναι καλά νέα. Όσο πιο φύλλα προσκύμενη είναι οι πρόεδροι μας ε, στη Ρωσία, τόσο καλύτερες είναι οι ευρωπαϊκές προοπτικές χώρας. Παράδοξο. Ε, χρειαζόμαστε πάντως ε, μια εκστρατεία ενημέρωσης της κοινή γνώμης ε, στην Ουκρανία για να του εξηγήσουμε στους πολίτες τι είδους ωφέλη θα αποκομίσουν. Παραδείγματο χάρη κατάργηση υποχρέωση θεωρήσεων και στη συνέχεια πραγματικές αλλαγές κράτους, δικαιο, δικαστικό σύστημα, τήρηση των πολιτικών ελευθεριών, νέα εισαγγελία, αντιμετώπιση της διαφθοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε Ευχαριστούμε ε, την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Τελωνιακή Ένωση. Hm. Η Ουκρανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παίξει ένα παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Ε, από τη μία πλευρά να υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη να αποπειραθεί να διαπραγματευθεί κάποιου είδους σχέση με την Τελωνιακή Ένωση. Διότι ε, το βασικό γκρόπ ψηφοφόρων του Προέδρου ε, είναι υπέρ των Ρώσων και αν κάνει οτιδήποτε διαφορετικό θα χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων του. Πρέπει λοιπόν αυτό να το συνυπολογίσουμε και να το έχουμε κατά νου. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε την υπογραφή της συμφωνίας και χρειαζόμαστε επίσης ε, ίσους όρους ανταγωνισμού με την Ρωσική Ομοσπονδία στις σχέσεις μας εφ' εξής. Όχι να επαν, να επαναπροσδιορίσουμε τις υφιστάμενες σχέσεις. Χρειαζόμαστε νέες σχέσεις. Ο Ρώσος ο πρόεδρος και η Ρωσία θα πρέπει να σέβονται το ότι η Ουκρανία είναι κυρίαρχο κράτος και γι' αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, παρακινήσαμε την ε, Ουκρανική κυβέρνηση και την Τιμοσέγκο και την Εισαγγελία και τι εκλογέ τα τρία αυτά ζητήματα, να τα προωθήσει και να τηρηθούν αυτά τα κριτήρια. Ευχαριστούμε, κύριο Σκλίτσκο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σα. Εν απαντήθηκαν από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Γιατσένιουκ. Να επιβεβαιώσω λοιπόν ότι σήμερα το θέμα είναι θα υπάρξει η Τελειονιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλειονότητα των Ουκρανών προτιμούν την ε, σύσφυξη σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι θα ωφεληθούν από αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι τα τρία τέταρτα των Ουκρανών δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ εκτός Ουκρανίας. Οπότε τις ευρωπαϊκές αξίες τις γνωρίζουν μόνο θεωρητικά. Βεβαίως, αν συγκρίνουμε το ΑΕΠ, των δύο πλευρών το βιωτικό επίπεδο, η υγεία, η κατάρτιση. Είναι σαφές ποιος υπερισχύει. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί είναι υπέρ της σύναψης ε, συμφωνίας σύνδεσης με την Ένωση. Θέλουν να είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές. Η Ουκρανία βεβαίως γεωγραφικώς ανήκει στην Ευρώπη, ιστορικά είμαστε Ευρωπαίοι. Η νοοτροπία μας είναι ευρωπαϊκή, αλλά ως βιωτικό επίπεδο απέχουμε πολύ, γι' αυτό θέλουμε να ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ήδη αναφέρθηκαν πολλά παραδείγματα, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία σημείωσαν μεγάλες προόδους, αυτό είναι καλό πρότυπο για την Ουκρανία. Βεβαίως ε, είναι σημαντικά τα καθήκοντα ενώπιών μας, πολλά βήματα πρέπει ακόμη να γίνουν μέχρι το Βίλνιους Αλλά μπορούμε να το επιτύχουμε, να επιτύχουμε ό,τι περισσότερα μπορούμε εμείς ως αντιπολίτευση για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρέπει να τα τα στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια. Πέντε εκλογικές περιφέρειες Ε, σε πέντε εκλογικές περιφέρειες πρέπει να ξαναγίνουν αναπληρωματικές εκλογές γιατί υπάρχουν ε, αμφισβητήσεις και στο Κίεβο πρέπει να γίνει αυτό. Είναι καθήκον μας. Όπως είπα και στην εισαγωγή μας, αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Η χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί χώρα ευρωπαϊκού επίπεδου όταν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά μας για να απελευθερωθεί η Γιούλια Τιμοσέγκα. Ε, είναι μεγάλο θέμα η διαφθορά. Πρέπει να καταπολεμηθεί, να υπάρξουν ε, μεταρρυθμίσεις. Και τέλος, είμαι πεισμένος ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται η Ουκρανία να είναι σταθερή χώρα οικονομικά και πολιτικά γιατί αν, υπάρξει, ε, αν υπάρξουν ε, ταραχές σε αυτή τη χώρα θα υπάρξει ε, θα είναι μεταδοτικό το φαινόμενο. Θα τα επιτύχουμε όλα αυτά μόνο προσεγγίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης. Είναι πρωταρχική σημασία για την Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Για αυτό το στόχο. Ως αντιπολίτευση κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι εξαρτάται από εμά. Είναι το όνειρό μας, είναι ο στόχος μας, θέλουμε να τον επιτύχουμε. Έχετε παρατήρηση για τον ε, G20 ναι, αναφέρεται το G20 και έχω να υπενθυμίσω ότι η προηγούμενη G8 ήταν G7 συν 1 και το G20 είναι 19 συν 1. Μετά το Snowden, μετά τη Συρία, μετά την Ουκρανία. Ας παραμείνουμε λοιπόν οι υπόλοιποι ενωμένοι για να έχουμε επιτυχία Νομίζω ότι η G20 από εμά εξαρτάται τι κατάληξη θα έχει η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε ενωμένοι. Εν τη ενώση η ισχύ και να επιδείξουμε θέληση να υπογράψουμε τη συμφωνία σύνδεση. Ε, Πρόεδρο, ούτω ή άλλω πληρώνει το φαγητό κύριο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είχαμε για να γίνει αυτή τη συζήτηση. Ε, Μπορούμε λοιπόν ε, να ε, έχουμε και να επανέχουμε αυτό το θέμα σε μιλήσια διάταξη ε, μέχρι τη Βίλνα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.